λοιπόν τα πρακτικά. Χθες λοιπόν ο πρόεδρος ανακοίνωσε μια ερμηνεία του κανόνα 202 παράγραφος 5 ε, που έχει προταθεί από την Επιτροπή για τα ε, σταγματικά θέματα. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανόνα 211 ε, αφού δεν είχαμε καμία αντίρρηση για αυτή την ερμηνεία εγκρίνεται. Έχουμε την πρώτη ανακοίνωση